Κύριοι, περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα έχουμε την εκλογή του διαμεσολαβητή ή της διαμεσολαβητού. Να επισημάνω το εξή. Θέλω την προσοχή σας λίγο γιατί πρέπει να προσπαθήσουμε να δείξουμε στον κόσμο πως είμαστε ένα τεχνολογικά προηγμένο κοινοβούλιο και άρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έχω, σας έχει δοθεί δύο φορές ε, οι οδηγίες χρήσης ε, του μηχανήματος, μία γραπτός και μία στο email σας. Παρ' όλα αυτά θα τις διαβάσω. Όταν ανοίξει η ψηφοφορία θα φανεί στην οθόνη σας μία παρουσίαση σαν αυτή που βλέπετε στις εικόνες που σας έχουμε μοιράσει. Εκεί πέρα στην οθόνη αναφέρεται το θέμα, δηλαδή εδώ πέρα στην περίπτωσή μας εκλογή του Διαμεσολαβητή. Και μετά βλέπετε τον κατάλογο των υποψηφίων. και τον αριθμό των ψήφων που είναι μία στην περίπτωσή μας. Μπορείτε να ψηφίσετε μία φορά. Δεν υπάρχει λίστα εδώ πέρα. Σημειώστε λοιπόν το όνομα του υποψηφίου ή της ε, υποψηφίας που θέλετε να ψηφίσετε με το μπλε κουμπί που υπάρχει κάτω δεξιά στην ε, συσκευή της ε, ψηφοφορίας Μπορείτε να πάτε πάνω και κάτω στον κατάλογο, να κινηθείτε στα ονόματα. Μετά μπορείτε να ψηφίσετε. Όταν φτάσετε στο όνομα που θέλετε, πιέζοντας το κουμπί ναι ή το κουμπί της αποχής. Δεν υπάρχει όχι. Είτε θα ψηφίσετε κάποιον είτε αποχή. Δεν υπάρχει αντίκη ψήφος. Επαναλαμβάνω. Όταν διαλέξετε με τον κέρσορα, τον δρομέα όπως λέγεται, το όνομα το οποίο θέλετε, μπορείτε να ψηφίσετε είτε ναι είτε αποχή. Μετά θα εμφανιστεί ένα αστεράκι δίπλα στο όνομα. Δηλαδή θα είναι το όνομα π.χ. Πλάσιντο Ντομίνγκο με αστεράκι. Αλλά μπορείτε να πατήσετε και να φύγει το αστεράκι αν θέλετε ε, να είναι μυστική η ψήφο σας. Με το μπλε κουμπί πάλι με το οποίο θα διαλέξετε υποψήφιο. Εάν το πατήσετε δεν θα φαίνεται το αστεράκι και κανείς δεν θα βλέπει ποιον ψηφίσατε. Νομίζω πως είναι τα πράγματα απλά. Ρωτάω λοιπόν, Υπάρχει κάποιος που δεν έχει καταλάβει τη διαδικασία και θέλει να ρωτήσει κάτι. Ωραιότατα. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, δεν είναι σωστό να βάλουμε τον Λουτσιάνο Παβαρότη ε, ως παράδειγμα, να δώσουμε τον Λουτσιάνο Παβαρότη παράδειγμα, δεν έχει αποβιώσει ο άνθρωπος. Οκ. Μάλιστα. Ε, τίποτα άλλο για το μηχάνημα έχετε να πείτε. Έχετε καταλάβει τη διαδικασία, ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Θα εμφανιστούν λοιπόν ονόματα και μπορείτε να επιλέξετε όπως το είπαμε. Και έχει τον εξής ε, στόχο. Σας διαβάζω από το άρθρο 204 παράγραφος 6. πρέπει πριν από την ε, ψηφοφορία να διασφαλίσει ο πρόεδρος πως είναι παρόντες τουλάχιστον οι μισοί βουλευτές. Εγώ θεωρώ πως είναι παρόντες αλλά πρέπει να το επαληθεύσουμε. Μπορείτε να ε, επιλέξετε μεταξύ του κυρίου Γκούσταφ Κλίντ, Αμεντέο Μοντιλιάνη, ο Γκούστ Ρενουάρ, Βίνσεντ Φανχόχ. Ε, ομολογώ πως βεβαίως έχουν όλοι ε, δυστυχώς ε, αποδημήσει. Ξεκινά λοιπόν η δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε ανάβει το μπλε λαμπάκι. Ψήφισαν όλοι λοιπόν. Πέρας της ε, ψηφοφορία. 617 ψήφισαν. Ογδόντα εννέα αποχές. Η ε, η απαρτία είναι 309. Ναι. Κανένα ζωγράφος δεν, δεν επέτυχε πλειοψηφία. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ε, κανονική ψηφοφορία. Κάνουμε ένα διάλειμμα για να προετοιμαστεί το σύστημα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις ε, ψηφ, με τις υποψηφιότητες. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Άλεξ Μπρένιγκ Μάιερ, τον κύριο Μάρκους Γέγκερ, την κυρία Ρία Ωμεν Ρόιτεν, την κυρία Έμιλι Οράιλι, την κυρία Ντάγμα Ροτμπέρεντ και τον κύριο Φραντσέσκο Σπερόνι που έχουν υποβάλει ψηφιότητες οι οποίες έχουν εξεταστεί και έχουν γίνει δεκτές. Λοιπόν, Άρχεται η ψηφοφορία. Haben alle... Ψήφισαν όλοι. Ξαναρωτάω, ψήφισαν όλοι. Ρωτάω για τρίτη φορά. Ψήφισαν όλοι. Ναι, οπότε πέρας της ε, ψηφοφορίας. Ψήφισαν 635, 78 αποχές, άρα η πλειοψηφία είναι 318 ψήφι, κανείς δεν επέτυχε την πλειοψηφία. Πρέπει να περάσουμε λοιπόν σε δεύτερο γύρο. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν έκανα λάθος. 713 ε, ψήφισαν. Οπότε επειδή δεν είχαμε εκλογή με την πρώτη ψηφοφορία. Αύριο θα έχουμε τον δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Ροτ Μπέρεντ για την ε, αλλαγή του κανονισμού των βλεφτών. Ε, υπαλλήλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπλοκ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεκτό. Μπλοκ 2. Άρα καταπίπτει. Όπως επίσης ε, και η ε, τροπολογία. Περνάμε τώρα στην ε, τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν. Παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Περνάμε τώρα στην πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. εγκρίνεται η έκθεση. Ο Επίτροπος ο κύριος Ζεύκοβιτς ε, ζητάει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποφεληθώ για να ευχαριστήσω εσά προσωπικά ιδιαίτερω, κύριε Πρόεδρε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ισχυρή υποστήριξη που δείξατε σε αυτέ τι δύσκολε διαπραγματεύσει. Χωρί την δική σα ε, προσωπική εμπλοκή ε, και ε, ε, δεν θα ήταν δυνατή αυτή η επιτυχία. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω την κυνησυγήτρια, την κυρία Ροτ Μπέρεντ και τους κοιόδης ηγητές Μπαλτάσαρ και Λίχτεμπεργκερ, Εξτρεμ Κάρι, Μαστόκα σπερόνι, γιατί συνεργάστηκαν, εργάστηκαν πολύ σκληρά και υπό χρονική πίεση. Χαίρομαι για τη σημερινή ψηφοφορία διότι εγκρίναμε ε, του, τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση και την διοικητική μεταρρύθμιση ε, που είχε προταθεί. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζεται με του Ευρωπαίου πολίτε. Ε, ενισχύει ε, ε, την εξοικονόμηση πόρων. Είναι μια πολύ καλή απόφαση και για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θα εξακολουθούν να μπορούμε να προσλαμβάνουμε τα ικανά στελέχη που χρειαζόμαστε και είναι σαφές και πάλι ότι η εργασία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δείχνει απλώς προσήλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποδεικνύει και ικανότητες ε, υψηλού επίπεδου ε, για να ξεπεράσει κανείς ε, δύσκολες δοκιμασίες. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να τελειώσω λέγοντας ότι πιστεύω πως μέσω, αυτής της, μέσω αυτού του εξυγχρονισμού η Ευρωπαϊκή Δημοσιοδιοίκηση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση και τις μελλοντικές προκλήσεις ε, εργαζόμενοι σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μιας Ευρώπης που θα είναι πιο ισχυρή ε, μετά την κρίση από όταν πριν από αυτήν. Ah, mi Να σα ανακοινώσω ότι από την ε, Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά, Πράσινη Ευρωπαϊκή Αριστερά, το αίτημα από τον κύριο Γκουλιάνη, την, τον ορισμό του κύριου κύριο Γκουλιάνη ω μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών. Δεν υπάρχουν παρατηρήσει, εγκρίνεται η τοποθέτηση. Πρώτο θέμα της κυρίας Μεζάρος